Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία τεσσάρων μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου των Σεϊχελών και δύο ψηλά ισταμένων του Κοινοβουλίου ε, και της αντιπροσωπείας ηγείται ο κύριος Βέιβεν Βίλιαμ. Βρίσκονται εδώ αυτή την εβδομάδα για να συμμετέχουν σε μία επίσκεψη τεσσάρων ημερών κατόπιν προσκλήσεως ε, του Γραφείου για την Προαγωγή της κοινοβουλευτική Δημοκρατίας. Ελπίζουμε η επίσκεψή σα αγαπητοί φίλοι να είναι επικοδομητική και ξέρουμε ότι θα παρακολουθήσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση του κυρίου Καντέκ για τη συμφωνία εταιρική σχέση ε, στην Αλληλεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σεχελών, η οποία θα ψηφιστεί αύριο. Σας ζητούμε στην επόμενη επίσκεψή σας να φέρετε και λίγο ήλιο για τις Βρυξέλλες.